Βλέπω ότι η κυρία Κρέιτον δεν έχει έρθει ακόμα και γι' αυτό θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπαρόζο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, τακτικά επισύρω την προσοχή σας στην έλλειψη